Η διάσκεψη των Προέδρων στη σημερινή της συνεδρίασης άμυ του παραρτήματος 16ου του Καρονισμού Λειτουργίας του Κοινοβουλίου ε, όρισε ότι ολοκληρώθηκε η ακρόαση του υποψηφίου επιτρόπου του Ηνωμένου Βασιλείου ε, και ως εκ τούτου προτείνει στην έγκριση της Ολομέλειας τη σχετική υποψηφιότητα. Προτείνω λοιπόν δυνάμει του άρθρου 152 παράγραφος 2 να περιληφθεί στην ημερήσια διάταξη των σημερινών μας ψηφοφοριών η έγκριση του, ε, της υποψηφιότητας του υποψηφίου επιτρόπου εκ μέρους του Βασιλείου. Υπάρχουν αντιρρήσεις παρακαλώ. Όχι. Και θα λάβει χώρα αμέσως η ψηφοφορία αυτή.